εξυγίαση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Η χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε μια καλύτερη ρύθμιση των διαφόρων χρηματοπιστωτικών παραγόγων και αυτό είναι το τελευταίο σημείο του, ε, ρυθμιστικού, του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Ε, θα ήθελα λοιπόν να παρατηρήσω το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουν ύψη την προτεραιότητα σε αυτό το θέμα στην επόμενη θητεία για να προστατεύσουμε τους επενδυτές και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα γενικώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, ε, τους τωρινούς και τους μελλοντικούς ε, ε, για τη συνεργασία τους και τη συνεργασία που είχαμε την τελευταία δεκαετία σε όλα τα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς που με απασχόλησαν. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Thank you. Και εμείς ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφε. Λοιπόν, ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφορία. η έκθεση Fox ε, για τους Ευρωπαίους Παρόχους Υπηρεσιών, μία και μόνο ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Κλείνει και αυτό το θέμα. Η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Έκθεση Ναχτεγκάλ ε, πρόκειται για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Ολοκληρώθηκε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έκθεση Κοντσολίνο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξης και Ταμείο Συνοχής. Ψηφίζουμε για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ μονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Η πρόταση απορρίφθηκε. Οι τροπολογίε των αρμόδιων επιτροπών ε, συλλήβδην όλε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. η τροπολογία τη αρμόδια επιτροπή, τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές ε, δεκτή, δεύτερη με ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η 18 σε δύο τμήματα, το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 19 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Τρίτο τμήμα με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 20 μονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η 41 σε δύο τμήματα, πρώτο, τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα, πάντα ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η 43 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία δεκτή. Η 59 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 60 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 66 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 67 υπέρ. 67 ηλεκτρονική επαλήθευση για την 67 παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή με πολύ μεγάλη ψηφοφορία. Η 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 82 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή 92 υπέρ κατά αποχές δεκτή 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή 98 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ έκλεισε η ψηφοφορία δεκτή 101 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ονομαστική κλίση ψηφίζουμε έκλεισε η ψηφοφορία Δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 102. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή η 106 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 225 υπέρ κατά αποχές δεκτή, απορρίπτεται, 226 ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 2.27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. 2.28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.12 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 229 υπέρ κατά αποχές δεκ, απορρίπτεται 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 231 καταπίπτει 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή η 2.33 καταπίπτει, η 2.34 ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε, έκκληση ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία 2-2, 2-0-2 0 κατά αποχές απορρίπτεται. 2-35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 196 και 203 μονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 71, 72, 73 υπέρ, κατά, αποχές, ε, δεκτές, 236 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 197 και 204 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Η έκκληση ψηφοφορία απορρίπτεται. 74, 75, 76 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 237 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 198 και 205 με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. απορρίπτονται 77, 78, 79 υπέρ, κατά, αποχές, ε, δεκτές. 2.38 ε, ονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. απορρίπτονται οι 83 και 191 υπέρ κατά αποχές δεκτές 84 και 192 υπέρ κατά αποχές δεκτές 193 υπέρ κατά αποχές δεκτή καταπίπτουν οι 85 και 86 239 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 87 και 194 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτές. 206 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Οι 2.40 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 2.41 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. απορρίπτεται και αυτή. 2.07 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.42D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.43 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Η 94, 95, 96, 97 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνονται δεκτές. Οι 2.13 καταπίπτει, οι 2.44D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 99 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε παρακαλώ, έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε, έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Καταπίπτει 208. Όχι, δεν καταπίπτει 208. Άρα ποιος είναι υπέρ της 208. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 185. Όχι, ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 208. Ψηφίζουμε ε, για τη 208. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η 185. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην 105 τμήματα, όλα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Δεύτερο. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πέμπτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 188, 199, 209, όχι, καταπίπτουν, καταπίπτουν όλοι, όπως και οι 214, πάμε στην 103D και 245D με ονομαστική κλίση, ε, ψηφίζουμε <laughs> έκκληση ψηφορία. Δεκτή. 186, ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε. έκκληση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 246D, ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 189, ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 108 ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. 2.47 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 2.48 δι ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.15 και 2.16 καταπίπτουν. Πάμε στη 2.17. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 195 και 201 μονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. απορρίπτονται. 11 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. 190 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 190. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Καταπίπτωση εκ τούτου 13, 14. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή καταπίπτει 2.19 187 διακόπτει ο πρόεδρος α, καταπίπτει και 187 Πάμε στην 15, ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε για την 15, έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. 2.20, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 223 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ έκλειση ψηφοφορία 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.24 ε, καταπίπτει. Ως εκ τούτου ψηφίζουμε για την πρόταση Επιτροπής με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Έγινε δεκτή η πρόταση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε. Έκθεση Ντάλι, πρότυπα επιδόσεων για, επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Ε, ψηφίζουμε, μονομαστική κλίση, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Δήλωση της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έκθεση ΡΙΣ, μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Ψηφίζουμε για την προσωρινή συμφωνία ε, με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε, έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Γίνεται δεκτή η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πάμε στην έκθεση Τουρκάνου προϊόντα λίπανσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε για την προσωρινή συμφωνία. Ψηφίζουμε μονομαστική κλίση παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ε, έκθεση Ατζέα, προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνου που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντε. Η συγγήτρια θέλει να λάβει το λόγο. Συγγνώμη, είναι δικαίωμα αυτό τη εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Με την τελική ψηφοφορία για αυτή την οδηγία σταθεροποιούμε το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πάρα πολύ ψηλές φιλόδοξες ε, ε, απαιτήσει και μπορέσαμε να εντάξουμε πάνω από 39 καρκινογόνες ουσίες ε, και αυτό θα πειράσει πολλά εκατομμύρια ανθρώπων και εργαζομένων κατά τα επόμενα έτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την Μαρίτα Ούστο κυρίω, ε, τον Κλόντ Ρολέν και άλλους από την Επιτροπή Απασχόλησης που μαζί με μένα ήταν οι συγητές στις δύο προηγούμενες οδηγίες. Να ευχαριστήσω και όλους τους και συγητές, όλους εκείνους που συμμετείχαν στην Επιτροπή μας γιατί κατέδειξαν ότι αυτό το Κοινοβούλιο πραγματικά μπορεί να έχει πολύ φιλόδοξους στόχους όταν αποφασίζει αποφασίσει να προστατεύει τους πολίτες. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε για την προσωρινή συμφωνία με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή με συντριπτική πλειοψηφία συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο έκθεση Αγίου του και κανόνε για ορισμένε συνδυασμένε εμπορευματικέ μεταφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Η συγγήτρια θέλει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κυρία Αγιούτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα του ηγητές από όλε τι ομάδε, οι οποίοι κατά τη διάρκεια διαχείριση αυτή τη οδηγία επέδειξαν ιδιαίτερο πνεύμα συνεργασία. Το κείμενο εγκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από την Επιτροπή Μεταφορών και είναι ένα σημαντικό στοιχείο τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα για να υπάρξει αποσυμφόρηση στι ευρωπαϊκέ οδού, να υπάρξει μεταφορά σε άλλα μεταφορικά μέσα πιο φιλικά προ το περιβάλλον. Μπροστά λοιπόν στου Ευρωπαίου πολίτε που σήμερα περισσότερο από ποτέ ζητούν την προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντο, αυτό το Κοινοβούλιο τάσεται υπέρ μια ευελιξία στην κινητικότητα. Και αυτό είναι ευκταίο. Θέλω να ελπίζω ότι και σήμερα θα στηρίξει το κείμενο ακριβώς όπως το ενέκρινε η αρμόδια επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε τη συνάδελφο. Ψηφίζουμε για το σύνολο των τροπολογιών της αρμόδιας επιτροπής. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές, δεκτές. Ε, τροπολογία 89 απορρίπτεται, 84D υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 30 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή, καταπίπτουν 85 και 86, 85 με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ, έκλειση ψηφοφορία. και απορρίπτεται. Η 90D υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η, να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 90D. Ε, ψηφίσαμε παρακαλώ, έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 82 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 88 καταπίπτει ως εκ τούτου και 83 καταπίπτει γιατί ε, απορρίφθηκε 87 ως εκ τούτου ψηφίζουμε για το σύνολο της πρότασης με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ Έκλειση ψηφοφορία Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη ανάγνωση. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πάμε στην επόμενη ε, έκθεση. Μπαγέ και Ραγνέρ, δημοσίευση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματο από ορισμένε επιχειρήσει και υποκαταστήματα. Ψηφίζουμε μετά την πρώτη ανάγνωση. Ποιο είναι υπέρ των αποτελεσμάτων τη πρώτη ανάγνωση. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στου συνεισηγητέ. Έκθεση Νοβάκοφ και Κρέλ. Κοινέ διατάξει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλά, το Ταμείο Συνοχή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία. Ψηφίζουμε τα συμπεράσματα τη πρώτη ανάγνωση. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στου συνεισηγητέ. Αντίρρηση, σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφο 3 του κανονισμού, μέσω χρηματοδοτική στήριξη των για το άσυλο και την μετανάστευση. Ψηφίζουμε το ψήφισμα χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ε, μεγάλη πλειοψηφία, αλλά αν θέλετε οπωσδήποτε έλεγχο, κλείνει η ψηφοφορία. Ε, εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά, μεγάλη πλειοψηφία. Αντίρρηση με βάση το άρθρο 105 παράγραφο 3 του κανονισμού μέσω χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων. Ισχύει το ίδιο όπω και προηγουμένω. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 107 του κανονισμού γενετικώ τροποποιημένη σόγια, μόνο 87751. Ψηφίζουμε το ψήφισμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. εγκρίνεται. Αντίρρηση σύμφωνα με βάση 107 του κανονισμού για το γενικό στροποποιημένο ραβόσιτο. Ψηφίζουμε το ψήφισμα με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού για τις ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισεθυλεξιλίου Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού ορισμένες χρήσεις του φθελικού δισεθήλεξιλίου. Ψηφίζουμε ολόκληρο το ψήφισμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τριοξίδιο του χρωμίου. Με αντίρρηση με το, βάση το άρθρο 106 του κανονισμού. Παράγραφος 1 του αρχικού κειμένου. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικό έλεγχο Για το αρχικό κείμενο. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Απορρίπτεται οριακά. Δεύτερο. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικό έλεγχος για το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρο... Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. εγκρίνεται όντως. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την τροπολογία 3 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. J, ε, αιτιολογική σκέψη, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη S υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη V υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την προηγούμενη αιτιολογική σκέψη, την S, αν και νομίζω ότι είναι η ίδια διαφορά, άρχεται η ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται όντω. Β. Αιτιολογική σκέψη, αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη χ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη ζ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη A-Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη α σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Διαδικαστικό ζήτημα ο κύριος Καβαντά. Μία, Μία φιλοφρόνηση. Μια... Και έχετε ξεκινήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες α, ε, της ταχύτητας. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διερμηνείς που κατάφεραν να σας παρακολουθήσουν αυτή την ηλικιώδη ταχύτητα που μιλάτε. Ε, τους ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ τους Διερμήνης λέω για το καταπληκτικό τους έργο. Ολοκληρώνουμε με την έκθεση Μπενιφέη, κατάσταση μετά την Αραβική Άνοιξη, μελλοντικέ ενέργειε για την περιοχή τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Παράγραφο 7. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Παράγραφο 47. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Παράγραφο. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για το δεύτερο τμήμα τη 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 48 αρχικό κείμενο, ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια, εγκρίνεται και συγχαρητήρια και σε όλους τους συναδέλφους. Yes, <laughs> I think so. Riprendiamo l'ordine dei lavori, colleghi. L'ordine del giorno reca ora la reazione. Συνεχίζουμε, περνάμε στην έκθεση φαγιών για τον κατάλογο τρίτων χωρών, υπήκοοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών, υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Κωσυφοπαίδιο. Συνάδελφοι, πριν λοιπόν δώσω το λόγο στη συνάδελφό μας, την κυρία Φαγιών, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ή δυνατόν να βγείτε από την αίθουσα τη ολομέλεια, αν δεν θέλετε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, αλλά χωρί να κάνετε φασαρία για να δείξετε και τον απαραίτητο σεβασμό προ την εισηγήτρια. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ελπίζω να επικρατήσει ησυχία στην αίθουσα, γιατί το θέμα είναι ευαίσθητο και πολύ σημαντικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, Δείξτε σεβασμό προς την εισηγήτριά μας, την κυρία Τάνια Φαγιό. Ευχαριστώ και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι. Συζητάμε σήμερα άλλη μια, για άλλη μια φορά την απελευθέρωση θεωρήσεων για το κοσυφοπαίδιο. Είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ δύσκολο θέμα αυτό, γιατί το Κωσυφοπαίδιο είναι η τελευταία χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που ακόμη δεν έχει καταργήσει τις θεωρήσεις για ταξίδια ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω σε όλους ότι το Κωσυφοπαίδιο έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις για ένα καθεστώς ελεύθερο θεωρήσεων εδώ και καιρό. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε πράσινο φως για να έχει το Κωσυφοπαίδιο καθεστώ ελεύθερο θεωρήσεων εδώ και καιρό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το Κωσυφοπαίδιο εκπλήρωσε όλα τα κριτήρια. Και σα θυμίζω το Κωσυφοπαίδιο είχε περισσότερες προϋποθέσεις ε, από οποιαδήποτε άλλη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων. Τα δύο τελευταία λεπτά θέματα τα αντιμετώπισε το κοσυφοπέδιο πριν από λίγους μήνες. Το ένα ήταν να ε, επικυρώσει την ε, συνοριογραμμή με το ε, Μαυροβούνιο, δύσκολο θέμα, τα κατάφεραν. Και επίσης ε, καταπολέμησαν την ε, διαφθορά σε υψηλά πολιτικά πρόσωπα. Έτσι λοιπόν η θερμή μου σύσταση είναι αύριο να επιβεβαιώσω με την απελευθέρωση των θεωρήσεων για αυτή τη χώρα. Για να είμαι ειλικρινή, όλε οι άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων έχουν σήμερα καθεστώ ελεύθερο θεωρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που θα σταλεί στου πολίτε των χωρών υποένταξη. Δεν είναι σημαντικό μόνο για πολιτική και οικονομικά ε, ζητήματα, αλλά και για τη σχέση μεταξύ των λαών. Σήμερα το Κωσυφοπέδιο είναι η πιο απομονωμένη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια και μιλούμε για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Δεν θέλω να συζητήσω για άλλα θέματα που αφορούν το Κωσυφοπέδιο, γιατί πρέπει συγκεκριμένα να δούμε τι ε, εκπληρώνει το Κωσυφοπέδιο. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να ασκήσω κριτική στις κυβερνήσεις που δεν ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις τους και τις υποσχέσεις τους ότι όταν θα εκπληρώσει τα κριτήρια θα χορηγήσω με το καθεστώς αυτό. Από το Συμβούλιο δεν είναι κανείς εδώ. Παρόλο, παρόλα αυτά ρωτώ, γιατί δεν το έβαλαν στην ημερήσια διάταξη και πότε σχεδιάζουν να βάλουν το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Χάνουμε την αξιοπιστία μας η χώρα και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες και δυνάμοι εγκληματίε δεν περιμένουν τις θεωρήσεις, ταξιδεύουν ελεύθερα. Αυτό που συζητούμε είναι ε, να μπορούν αυτοί που έχουν ανάγκη να ταξιδέψουν, με κάποιους περιορισμούς βέβαια έχει κάποιου περιορισμούς ε, το ταξίδι ελεύθερο θεώρηση και το ε, γνωρίζουν. Η εκστρατεία συνεχίζεται και πρέπει να ανταποκριθούμε στι υποσχέσει μα. Σα θυμίζω και άλλε περιπτώσει. όπου ανταποκριθήκαμε και δώσαμε στην Ουκρανία τέτοιο καθεστώ εν μια νυχτή. Ήταν πολύ εύκολη η πολιτική απόφαση και τώρα οι Ευρωπαϊκέ κυβερνήσει μπλοκάρουν μια μικρή χώρα των Δυτικών Βαλκανίων χωρίς λόγο πραγματικό. Ε, καλό όλους, γιατί η θητεία μας ολοκληρώνεται, αύριο να επανεπιβεβαιώσουμε ε, την εντολή που μου εδόθη, δηλαδή ότι στηρίζομαι το καθεστώς ελεύθερο θεωρήσεων για το κοσυφοπαίδιο. Ε, το ξαναλέω, εξεπλήρωσε όλες τις προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναγνώρισε. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι εκείνες που σήμερα δεν αναλαμβάνουν δράση. Έχουμε πολλές περιπτώσεις ε, όπου οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπλοκάρουν τις αξιόπιστες ευρωπαϊκές μας πολιτικές και η πολιτική των θεωρήσεων είναι πραγματικά στην καρδιά των Ευρωπαίων. Είναι κάτι απτό και καταλαβαίνω την αγανάκτηση των ε, πολιτών του Κωσυφοπεδίου όταν νιώθουν ότι τους ζητούμε να κάνουν κάτι, το κάνουν και εμείς τώρα δεν ανταποκρινόμαστε. Εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, τώρα η μπάλα είναι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Αύριο θα ψηφίσουμε για την ε, εντολή και ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση, παρακαλώ ε, υποστηρίξτε την εκθέση αυτή γιατί ο λαός του Κωσυφοπεδίου μας παρακολουθεί με μεγάλες προσδοκίες και ελπίδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την αγαπητή συνάδελφο και ζητώ συγγνώμη για το γεγονό ότι στην αρχή, όταν αρχίσετε την παρέμβασή σα, υπήρχε έτσι κάποια φασαρία στην αίθουσα και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο. Παρακαλώ πολύ, κύριε Αβραμόπουλε. Γκράτσι, ε, κύριε Πρεζιντέντε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συζήτηση αυτή για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για το λαό του Κωσυφοπεδίου. Και θα ήθελα να εκφράσω και πάλι τις ευχαριστίες μου προς την εισηγήτρια, την κυρία Φαγιό, για την συνεχή της προσπάθεια, προσωπική δέσμευση και ε, όλες τις προσπάθειες που έκανε για να στηρίξει αυτή την έκθεση. Ήδη από το 2012, το διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με το Κωσυφοπαίδιο, βοηθώντας τις αρχές να τηρήσουν όλα τα κριτήρια του δικού χάρτη για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Και στην τελική μας έκθεση πρόοδου της 4 η Μαΐου του 2016 αναγνωρίσαμε ότι το Κωσυφοπαίδιο έκανε σημαντικά βήματα προς ένα καθεστώς ε, χωρίς θεωρήσεις. Και γι' αυτό προτείναμε την άρση της υποχρέωσης θεώρησης ε, διαβατηρίου για το λαό του Κωσυφοπεδίου ε, θεωρώντας ότι την ημέρα της ε, έγκρισης πρότασης από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Κωσυφοπέδιο θα έχει κυρώσει την οριοθέτηση των συνόρων με το Μαυροβούνιο και θα έχει σημειώσει πρόοδο στην πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Δύο χρόνια μετά, 19 Ιουλίου του 2018 και μετά τις απαραίτητες προσπάθειες και την πρόοδο που έχει στελεστεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το κοσυφοπαίδιο έχει τηρήσει όλες τις προϋποθέσεις για το νοδικό χάρτη για την άρση των θεωρήσεων και τις δύο εκκρεμείς προϋποθέσεις που προανέφερα. Ως εκ τούτου, ζητήσαμε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν την πρότασή μας. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που επιφύλαξε στην πρότασή μας. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η σύναψη της συμφωνίας οριοθέτηση των συνόρων με το Μαυροβούνιο είναι ένα τεράστιο βήμα πρόοδου και καθόλου εύκολο και δεδομένο. Παρόλο που το θέμα είναι πολιτικώς ευαίσθητο και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Κάποιες χώρες εξέφρασαν ε, ε, ανησυχίες για τις μεταναστευτικούς κινδύνους από τους κατοίκους του Κωσυφοπεδίου και την ανάγκη να διδαχθούμε από το παρελθόν. Έχω επίγνωση αυτού του προβληματισμού και θεωρώ ότι είναι ευνόητες ε, και εύλογες οι ανησυχίες. Αλλά επίγνωση έχει και το Κωσυφοπέδιο και συνεργάζεται μαζί μας και έχει άμεσες επαφές με τα ενδιαφερόμενα κρατημέλη για να μετριάσει τους κινδύνους. και στο παρελθόν ενθαρρύναμε τις αρχές του Κωσυφοπεδίου και θα το κάνουμε και στη συνέχεια για να εφαρμόσουν όλα, όλους τους γνώμονες. Επίσης να συνεχίσουν και να ενισχύσουν το πλαίσιο πάταξης διαφθοράς και φυσικά να συνεχίσουν το έργο τους για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Και επίσης επισημάνουμε την ανάγκη ε, σωστή επικοινωνία και ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει του δυνάμει του καθεστώτο απελευθέρωση θεωρήσεων. Άλλωστε, το Κωσυφοπέδιο είναι η μόνη χώρα εταίρο από τα Δυτικά Βαλκάνια που δεν επωφελείται από ε, διευκόλυνση θεωρήσεων. Και οι πολίτε του Κωσυφοπεδίου είναι οι μόνοι στην περιοχή που χρειάζονται θεώρηση διαβατηρίου για να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω δηλώσει επανειλημμένω ότι η απαλλαγή από τις θεωρήσεις ε, συνεπιφέρει δικαιώματα και υποχρεώσεις και οι αρχές του κοσυφοπεδίου το γνωρίζουν. Έκαναν το καθήκον τους και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους. Και ενθαρρύνω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καθίσουν στην ε, Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και να εγκρίνουν το συντομότερο δυνατό την πρόταση. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Επίτροπε. Εκ μέρους Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων τώρα το λόγο ο κύριος Σόλτες για ένα λεπτό. Βαλά. Ε, ευχαριστώ. Ως μόνιμος εισηγητής για το Κωσυφοπαίδιο στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την ΑΦΕΤ, θα ήθελα να πω ότι το Κωσυφοπαίδιο αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις. Πριν από ένα χρόνο ε, κυρώθηκε η συμφωνία για τα σύνορα με το Μαυροβούνιο και αυτό ήταν ένα επίτευγμα. Γιατί ε, έπρεπε να γίνει εσωτερική συνεννόηση και συμφωνία. Και αυτό ήταν το τελευταίο βήμα προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης από την, ε, τις θεωρήσεις. Επίσης, πρόοδος επιτελέστηκε στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος της διαφθοράς και η Ευρώπη διαβεβαίωσε ότι ε, όλα τα βήματα είχαν γίνει και θα ανταποκρινόταν. Μετά όμως δεν ε, έγινε τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς στο Κοινοβούλιο δώσαμε το πράσινο φως για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Παρ' όλα αυτά όμως το σημείο αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Έχουμε δύο εταίρους. Ο ένας εταίρος ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και ο άλλος όχι. Εν προκειμένου ο δεύτερος εταίρος χάνει σε αξιοπιστία και υποχρεούμεθα ε, να προχωρήσουμε υπέρ των, του λαού του Κωσυφοπεδίου. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στα πολιτικά κόμματα εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ο κύριο Αντέμοφ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την έναρξη του διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κωσυφοπεδίου είχαμε τέσσερις εκθέσεις πρόοδου για το Κωσυφοπέδιο και το Μάιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις δύο προτάσεις της για το Κωσυφοπέδιο για την κύρωση της συμφωνίας της οριοθέτησης του συνόρου με το Μαυροβούνιο και την ανάγκη να, να συνεχίσει την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και την πάταξη τη διαφθορά. Συντρέχουν πια και οι δύο προποθέσει. Ε, εκπλήρωσε και τι δύο υποχρεώσει το Κωσυφοπέδιο, όπω προκύπτει από την έκθεση πρόοδου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2018. Επιπλέον, το Κωσυφοπέδιο χρειάστηκε να συμπληρώσει άλλα 95 κριτήρια και τα έχει ε, πραγματοποιήσει όλα. Οπότε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες της κοσοβάρικης κυβέρνησης ε, ήρθε επιτέλους η ώρα να δείξουμε στο λαό του Κωσυφοπεδίου, στους πολίτες του Κωσυφοπεδίου, ότι πραγματικά νοιαζόμαστε για αυτούς. Ενδιαφερόμαστε για τους φίλους μας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι εφόσον τηρήθηκαν οι υποσχέσεις, εφόσον υλοποιήθηκαν τα κριτήρια, θα κάνουμε και εμείς το καθήκον μας και θα ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες των Κωσοβάρων. Δηλαδή, θα επιτρέψουμε στο λαό του κοσυκοπαιδίου να ταξιδεύει ελεύθερα και χωρίς ανάγκη θεώρηση διαβατηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ακούσαμε, το Κωσυφοπαίδιο είναι η μόνη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που δεν επωφελείται από την απαλλαγή τη υποχρέωσης θεώρηση. Και φυσικά η απελευθέρωση των θεωρήσεων δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα. Θα σας υπενθυμίσω ότι πολύ ετούντες άσυλο από το κοσυφοπέδιο, ο αριθμός των ετούντων άσυλο από το κοσυφοπέδιο έχει μειωθεί δραστικά. Μάλιστα ξεκίνησε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης στο κοσιφοπέδιο για τις υποχρεώσεις που συνεπιφέρει ένα τέτοιο καθεστώς απελευθέρωσης θεωρήσεων. Επίσης έχει θεσπίσει και ένα νομοθετικό πλαίσιο η χώρα που καλύπτει όλες τις μορφές τρομοκρατίας και προβλέπει και κάποια εργαλεία διεθνώς για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των οργανωμένων εγκλήματος. Επίσης, το κοσυφοπαίδιο εκπλήρωσε όλες τις απαιτήσεις μας και για τις επιστροφές και για την επανένταξη των πολιτών, τη διαχείριση των συνόρων, την δημόσια τάξη και την ασφάλεια. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι θα πρέπει να υπερψηφίσουμε την απελευθέρωση των θεωρήσεων για το κοσυφοπαίδιο. Πολύ ωραία. Εκ μέρου ε, των Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Ζίπελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήδη πριν από περίπου τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το κοσοπέδιο να απαλλαγεί από την υποχρέωση για θεώρηση. Γιατί ήδη και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πεπισμένη ότι το κοσυφοπέδιο θα εκπληρώσει έγκαιρα και τις τελευταίες προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Το γεγονός ότι αυτό συνέβη, αυτό το επιβεβαίωσε η Κομισιόν ήδη τον προηγούμενο Ιούλιο. Και όμως παρόλα αυτά σήμερα εμείς δεν συμφωνούμε, δεν ψηφίζουμε μάλλον για το αποτέλεσμα ε, τριμερούς διαλόγου. Ε, Ακόμα λοιπόν καθυστερούμε και ορισμένα κράτη-μέλη μπλοκάρουν τις διαπραγματεύσεις. Αυτό απομονώνει το κοσφοπέδιο και καθυστερεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πώς θα εξηγήσουμε λοιπόν στους ανθρώπους στο κοσφοπέδιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά από το πουθενά βγάζει από το καπέλο της άλλες προϋποθέσεις τη στιγμή που η χώρα έχει ήδη καλύψει όλες τις προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Αυτή λοιπόν η στάση δεν συμβάλλει στο να ε, παραμείνει αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση στους Κωσοβάρους. Οι υποσχέσεις που δώσαμε εμείς στο κοσφοπέδιο πρέπει να τηρηθούν. Ναι, πράγματι, ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσοπέδιο ως κρατική οντότητα, ως κράτος. Όμως αυτό δεν είναι απαραίτητο για να δοθεί απελευθέρωση από τη θεώρηση. Δεν χρειάζεται να αναγνωρίσει κανείς το κράτος. Αρκεί να αναγνωρίσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία και τώρα είναι ασφαλή. Δεν μπορούμε πια να ε, κρατάμε το κοσμοπέδιο στο να περιμένει. Καλύπτονται οι προϋποθέσεις, η θέση του Κοινοβουλίου είναι απόλυτα σαφής και έχει φτάσει πια η στιγμή το Συμβούλιο που και πάλι λάμπει δια της απουσίας του να τοποθετηθεί έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να τηρήσει την υπόσχεσή της συνολικά, στο σύνολο των κρατών μελών. Ωραία. Τώρα, εκ μέρου ε, των συντοριτικών και μεταρρυθμιστών, ε, Βίστησεν, ε, παρακαλώ. Ο κύριος Βίστησεν. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλοί έγκυροι λόγοι που με κάνουν επιφυλακτικό σε σχέση με την απελευθέρωση και το κοσυφοπαίδιο. Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα μη ε, ασυρά χωρών δεν αναγνωρίζουν το Κωσυφοπαίδιο σαν εξάρτητο κράτος και αυτό δυσκολεύει το Συμβούλιο να αναλάβει δράση που, σε ένα θέμα που έχει μπλοκαριστεί. Ένα βασικό πρόβλημα για μένα και για το ECR είναι η εστίαση στη μονόπλευρη ε, απελευθέρωση των θεωρήσεων. Όταν πρόκειται περί του οργανωμένου εγκλήματος, Έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών προβλημάτων στα Δυτικά Βαλκάνια εν γέννη και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εύλογο να εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση της θεώρησης εν προκειμένου. Ε, Επίση, προσωπικά ανησυχώ πάρα πολύ βλέποντας την ε, ριζοσπαστικοποίηση που διαδίδεται όλο και περισσότερο στα Δυτικά Βαλκάνια. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και η υποχρέωση της θεώρησης είναι καλό για να φιλτράρουμε τον αριθμό των εισερχομένων στην Ένωση. Η Ένωση θα πρέπει να εστιάσει στις συμφωνίες επιστροφής, προκειμένου περί μεταναστών που πρέπει να επιστραφούν και όχι να απελευθερώνουμε τα καθεστώτα θεωρησέων. ο ομιλητή, ο κύριος Μιλινάρ, η κυρία Μιλινάρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Να ευχαριστήσω την Τάνια Φελιών, την εισηγήτρια και όλους τους κοιόδης καταρχήν. Έκαναν πολλές προσπάθειες. Το φάκελος ε, συνεχιζόταν την χάνει επεξεργασίας, ενώ η Κομισιόν είχε ήδη προτείνει την απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων ε, μεταφέροντάς το στον κατάλογο αυτών που είχαν δικαίωμα για σύντομη παραμονή. Τον περασμένο Ιούλιο ανακοινώθηκε ότι οι, δύο πιο σημαντικές προϋποθέσεις είχαν αρθεί. Καταρχήν κυρώθηκε από το Κωσυφοπαίδιο Συμφωνία για τα σύνορα με το Μαυροβούνιο και δεύτερον είχε ε, βελτιώσει τις επιδόσεις του στον τομέα της καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς. Το Σεπτέμβριο το Κοινοβούλιο ε, ψήφισε υπέρ των διοργανικών διαπραγματεύσεων και θα ψηφίσουμε ε, θετικά αύριο, ούτω ώστε να οριστικοποιηθεί το θέμα στην επόμενη θητεία. Το Πέδιο απομονώθηκε στα Βαλκάνια ε, για πάρα πολύ μεγάλο, υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Η απελευθέρωση των θεωρήσεων θα ήταν ένα δίκαιο βήμα προς τη χώρα αυτή. Ε, είναι ε, ε, πολλοί λόγοι. Θα διευκολυνθούν οι διαπροσωπικές επαφές, θα ανταλλαγούν, θα γίνουν ανταλλαγές σε πολλά επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό κλπ. Επίσης θα μπορέσει η Ένωση έτσι να προωθήσει περισσότερες μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η απαλλαγή μπορεί να ε, ε, ε, επηρεάσει και τον τομέα των υπηρεσιών. καλό να, αρχίσουν να αρχίσει η διαδικασία αυτή. Δεν υπάρχει πια λόγος να δυσκολεύουμε την είσοδο στο χώρο του Σέγγεν των πολιτών του κοσύφε Πεδίου. Πρασίνο, ε, η κυρία Βαλέρο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τότε που ανέκτησε την ανεξαρτησία του, το Κωσυφοπέδιο είχε αναγνωριστεί από 23 χώρες. Και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης δεν θεωρεί ότι η ανεξαρτησία του Κωσυφοπέδιου αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Και μάλιστα πέντε χώρε ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ρουμανία και η Σλοβακία δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το κοσυφοπαίδιο ως ανεξάρτητη χώρα. Οπότε δεν προβλέπεται εξαίρεση από το καθεστώ θεώρηση. Παρ' όλα αυτά, το κωσυφοπαίδιο έχει εκπληρώσει και τα 95 κριτήρια. Τώρα εναπομένει σε εμά να κάνουμε το καθήκον μας. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε αξιοκρατικά την απόφασή μας και όχι να κατευθυνόμαστε από πολιτικά κίνητρα ή πολιτικά παζαρέματα. Και μάλιστα χώρες που δεν αναγνώρισαν το κοσυφοπαίδιο ψήφισαν υπέρ της απελευθέρωσης της ε, Ειδικευμένες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Εμείς οι πράσινοι στηρίζουμε πάντως τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ και τώρα εκ μέρους της ΓΚΟΕ το λόγο έχει η κυρία Βερζιά. Για δύο λεπτά. Μαρή Κριστίν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Το Κωσυφοπέδιο έχει λιγότερο από 2 εκατομμύρια κατοίκους. Έχει ε, βουτυχθεί στο αίμα από τον πόλεμο με 13.000 νεκρούς και είναι η μόνη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που δεν υποφελείται από απελευθέρωση των θεωρήσεων. Βραχίας διαμονής βέβαια γιατί είναι οι μόνες ε, θεωρήσεις που εμπίπτουν στην ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αλβανία έχει τέτοιο καθεστώς από το 2010, η Σερβία και το Μαυροβούνιο από το 2008. Το Κωσυφοπαίδιο είναι η μόνη χώρα απομονωμένη που δεν επωφελείται από την απαλλαγή των θεωρήσεων. Και μάλιστα έχει εκπληρώσει τα πιο λεπτομερή και πολυάριθμα κριτήρια από τι άλλε χώρε. Και το έχει κάνει. Και μάλιστα την νομοθετική τη πρόταση το 2016 την κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα ε, και ενώ με το Τόγκα και άγνωστα ε, νησιά, το Βανουάτου, ε, επισπεύδουμε τις εμπορικές μας συμφωνίες, και τις συμφωνίες απαλλαγής ε, θεωρήσεων, παρόλο που σχεδόν αποκλείεται να έρθουν ε, στην επικράτειά μας, ε, έχουμε επισπεύσει τις προσπάθειες. Ενώ για το κοσυφοπαίδιο δεν είμαστε αρκετά γρήγοροι. Για να μην μιλήσουμε για το ρόλο του αιτία και άλλων βάσεων δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πολλέ προσπάθειε και το Κωσυφοπέδιο επίση πολύ περισσότερο από ό,τι γειτονικέ χώρε. Μιλήσαμε για τη διαφθορά του ε, δικαστικού συστήματο, αλλά δεν είναι η μόνη χώρα που έχει τέτοια προβλήματα. Επίση, το 2016 είχαμε τη διαπραγματευτική εντολή και το 2018 επιβεβαιώσαμε και εμεί αυτή την εντολή. Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει την ε, διαπραγματευτική εντολή. Και επίση πέντε χώρε ακόμη δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπαίδιο. Η Γκουε είναι αναφαδόν υπέρ τη απελευθέρωση των θεωρήσεων και τη ελευθερία διακίνηση. Δεν θέλουμε καμία εξαίρεση για το κοσυφοπαίδιο και διάκριση σε σχέση με τι άλλε χώρε. Συμφωνώ με την εισηγητρία την κυρία Φαγιόν και την ευχαριστώ για την αιμονή που έχει δείξει. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και τώρα, εκ μέρου τη Ευρώπη των Εθνών και τη Ελευθερία, ο κύριο Ζήλστρα για 1,5 λεπτό. Ο κύριο Ζήλστρα, παρακαλώ, κύριε Ζήλστρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για λόγους ασαφής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χορηγήσει το καθεστώς απαλλαγής, αποθεωρήσει σε πολλές χώρες και στο κοσυφοπαίδιο τώρα. Το κοσυφοπαίδιο κήρυξε την ανεξαρτησία του που όμως δεν αναγνωρίστηκε από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν και προβλήματα με εγκληματικέ συμμορίες ε, από το κοσυφοπαίδιο που πάνε στην υπόλοιπη Ένωση. Μπορούν να σταματήσουν στα σύνορα, αλλά η Κομισιόν φαίνεται να μην το θέλει αυτό. Ε, δεν υπάρχει κράτος δικαίου ε, στο Κωσυφοπαίδιο και αυτό ε, επιβεβαιώθηκε κατά τις αποστολές. Ε. Υπάρχουν προβλήματα με τις ιερόδουλες, τα, τις συμμορίες, οι διοκτικές αρχές κάνουν ότι δεν βλέπουν. Υπάρχουν περιγραφές για την κατάσταση στο Κωσυφοπαίδιο μετά από αποστολές πέρσι ε, ε, ε, που περιγράφουν το κοσυφοπέδιο ως ένα καράβι με διαρροή, το οποίο θα βυθιστεί. Γιατί υπάρχει η υποχρέωση από τη δική μας την πλευρά. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι υπέρ. Εμείς θα ψηφίσουμε κατά. Το λόγο έχει για ένα λεπτό. Grazie, Presidente. Τα πλεονεκτήματα ε, για τους πολίτες μιας υποένταξη χώρας όπως είναι το κωσυφοπαίδιο από την απαλλαγή της υποχρεώσεως θεωρήσεως των διαβατηρίων είναι προφανή. όμως η εξασφάλιση αλλά και η διατήρηση αυτού του πλεονεκτήματος πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα της κυβερνήσεως της χώρας. προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση του κωσυφοπαιδίου παρά τις κάποιες προσπάθειες που έχει καταβάλει δεν έχει επιτύχει να εκπληρώσει τους περισσότερους από τους απαραίτητους όρους πέραν του γεγονότο ότι δεν έχει καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα έχει επιτρέψει να γίνει η χώρα καταφύγιο τρομοκρατών και δολοφόνων του isis. επιπλέον με την συμπεριφορά τη προκαλεί τι γειτονικέ χώρε. παραδείγματο χάρη βλέπουμε να υπάρχουν συνεχή συνοριακά επεισόδια με τη σερβία. επιπλέον επιβάλλει δασμού στα προϊόντα που έρχονται από τη σερβία. Επίση, μεθοδεύει την συνομοσπονδία με την αλβανία η οποία ω γνωστόν εγείρει επεκτατικές βλέψεις και εδαφικές ε, αξιώσεις επί του διαμερίσματος της υπήρου της ελλάδος. κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι αδιανόητο θεωρώ αυτή τη στιγμή να συζητούμε και για την αναγνώριση του κωσυφοπεδίου αλλά και για την ε, άρση του εμποδίου που προκύπτει από την θεώρηση